Ελπίσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι θα διεξάγουμε αυτή την εκστρατεία για τον εμβολιασμό γιατί αλλιώς αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι τζάπα η δουλειά μας. Δεν θα έχει οδηγήσει τίποτα. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ε, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε στις 12 και ε, το επόμενο θέμα είναι κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο. Πρώτη μιλήτρια κυρία Ματσόνη. Η Ερμήνια. Yes, it's okay. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα η ερώτηση που έχουμε υποβάλει ως Επιτροπή των Αναφορών ε, αποδεικνύει πως ε, η δική μας ε, η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη για την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στο θέμα το οποίο ετέθη από την Ισπανική Ομοσπονδία Παραγωγών και Εξαγωγέων Οποροκυπευτικών Ουλουδιών και Ζώντων Φυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει τη δική της την προσοχή στο γεγονός ε, ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που φέρουν την ευθύνη στον καθορισμό ε, ορισμού τιμών. Πρέπει όμως ε, να ληφθεί υπόψη αυτό που ελέγχθη από την Επιτροπή Αναφορών. Δηλαδή η καταγγελία όσον αφορά τις παρατυπίες στην εισαγωγή ε, της ντομάτας και άλλων οποροκυπευτικών από το Μαρόκο. Αυτή λοιπόν η παρατυπία ετέθη ήδη πριν από κάποιο καιρό, πριν από ένα χρόνο περίπου, από την Όλαφ, από τον Οργανισμό Ελέγχου, η οποία Όλαφ πράγματι διαπίστωσε ότι υπάρχει κάποια παρατυπία η οποία βασίζεται στον μηχανισμό εξαίρεσης ο οποίος πρέπει τον κανονισμό 32-34 που προβλέπει τρεις διαφορετικούς υπολογισμούς της τιμής εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση αυτής της μεθόδου προσφέρει στους αγωγείς τη δυνατότητα να μην καταβάλουν τους δασμούς και αυτό οδηγεί σε ανομαλίες στην αγορά. Κατ' ουσίαν το γεγονός αυτό οδηγεί ε, στη μείωση του εισοδήματο ε, των ε, παραγωγών αλλά και των εξαγωγών αγωγέων ντομάτα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ άλλων στις χώρες Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται μια νέα διμερή συμφωνία με το Μαρόκο. Στη συμφωνία αυτή για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ανησυχητικά στοιχεία που σας ανέφερα. Και φαίνεται ότι τελικά ε, θα εφαρμόζεται ε, εισαγωγή ντομάτας από το Μαρόκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία εισαγωγή όμως που δεν ε, διέπεται από τους δικούς μας τους κανονισμούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, ένα θέμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του ή αν θέλετε ε, φύγει ε, ένα πολύ λεπτό σημείο που προέκυψε ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό το σημείο είναι οι ε, μεταναστευτικές ροές. Έχουμε όλους αυτούς τους πολίτες που έρχονται από χώρες όπως είναι και το Μαρόκο, δηλαδή από χώρες της Βόρειας Αφρικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι μεταναστευτικές ροές δημιουργούν προβλήματα στις χώρες μας, προβλήματα και στη γεωργία. Εμείς λοιπόν έχουμε τεράστια δυσκολία να δεχθούμε τους μετανάστες αυτές, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ιταλία κυρίως έχουμε τεράστια δυσκολία να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ελπίδα ζωής. Γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής των δικών μας των χωρών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και προκύπτουν πολύ μεγάλες ζημιές. Και θα ήθελα να γνωρίζω τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Commissioner, Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέψετε θα προσπαθήσω να απαντήσω στα αρκετά ερωτήματα που έθεσε που έχουν τεθεί με την αναφορά και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαρτσόνη, η οποία υπέβαλε την προφορική αυτή ερώτηση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σα ε, καθησυχάσω. Η Επιτροπή παρακολουθεί την ποσότητα εισαγόμενων τοματών από το Μαρόκο πολύ προσεκτικά με ένα σύστημα διασταύρωση βάσει τη δήλωση ε, των ποσοτών που εισάγονται ε, και των ημερήσιων ε, εισαγωγών όπως αυτές καταγράφονται από τις τελωνιακές αρχές. Μέχρι σήμερα η Κομισιόν δεν έχει καμία απόδειξη συστηματικής απάτης ή αστοχίας του συστήματος που έχει σε λειτουργία. Έχουμε πληροφορία για μία περίπτωση, θα επανέλθω σε αυτή λίγο αργότερα. Και αφορά το έτος 2007, όπου η Όλαφ πράγματι τόνισε ότι το σύστημα ως είχε θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες καιροσκοπικές συμπεριφορές αλλά όχι πάντα και σε παρατυπίες. Σε ό,τι αφορά την ε, τιμή εισόδου ή την ίσπραξη κάποιων δασμών, πράγματι αυτά αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών. Μια άλλη πτυχή που είναι αρκετά σημαντική για το θέμα αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο, δηλαδή γύρω στις Ντόχα οποίο και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Οποιαδήποτε αλλαγή λοιπόν στην τιμή εισόδου και στο πώ εφαρμόζεται θα μπορούσε να περάσει αρνητικά τα μέχρι τούδα αποτελέσματα. Η νέα δημορή συμφωνία με το Μαρόκο προστατεύει ε, τα συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων εμπόρων και καταναλωτών και βέβαια προβλέπει και μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη διαφάνεια τα δεδομένα εμπορία οπωροκυπευτικών ποσοτική αύξηση έχει περιοριστεί στους 52.000 τόνους. Είναι προοδευτική και θα γίνει μέσα σε τέσσερα έτη εμπόριας. Άρα προστατεύεται η παραδοσιακή εισαγωγή και προμήθεια και φοδίσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και για την αλλαγή τιμών εισόδου πρέπει να γίνουν σεβαστέ οι σχετικέ ε, διεθνεί συμφωνίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο κανονισμό εφαρμόζεται σωστά εξού και ξεκίνησε έρευνα μέσω τη Όλαφ και νομίζω ότι για αυτήν την περίπτωση έκανε λόγο η κυρία Ματσόνη. Σε ό,τι αφορά παρατυπίες από μη ορθή ερμηνεία των ε, κανόνων εφαρμογή, είναι ευθύνη των εθνικών κρατών να παρακολουθούν τα αποτελέσματα η ανάκτηση είναι σε εξέλιξη, αλλά η δημοσίευση των δεδομένων αποτελεί, επαναλαμβάνω, αρμοδιότητα των αρμοδίων τελωνιακών αρχών. Σε ό,τι αφορά τώρα την οργάνωση της επιτήρησης, ένα από τα θέματα τα οποία τέθησαν από την κυρία Ματσόνη. Εδώ πρέπει να πω ότι η Επιτροπή, όπως είπα, παρακολουθεί τις εισαγωγές τομάτας από το ε, Μαρόκο με ένα σύστημα ταυρούμενου ελέγχου. Επί εβδομαδίας βάσεως γίνεται αυτή η παρακολούθηση και τα δεδομένα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα τα οποία παρέχουν οι εθνικές τελωνιακές αρχές και τα δεδομένα της Eurostat. Άρα νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές ακριβείς πληροφορίες, οπότε ε, αν υπάρξουν συστηματικές απάτες ή παρατυπίες, αυτές θα εντοπιστούν και αμέσως θα αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρία ερανθ γκαρθη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών για το έργο που έκανε μετά την καταγγελία ε, της ΘΕΠΕΞ, e δηλαδή τη Ισπανική Ομοσπονδία Παραγωγών και Εξαγωγών Οποροκυπευτικών βάσει τη έκθεση που δημοσίευσε η Όλαφ το 2007. Νομίζω τα συμπεράσματα τη έκθεση είναι ξεκάθαρα και δικαιολογούν άκρο αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχε κάνει εδώ και καιρό η Κομισιόν για να ευκρινίσει αυτό το σύστημα υπολογισμού των τιμών ε, εισόδηδε ό,τι αφορά τον τομέα τη ε, ντομάτα. Υπήρξαν ενδεχομένω ε, κάποιε παγίδε ε, λόγω του υπολογισμού τη τιμή εσόδου. Όχι μόνο δεν έλειψαν αυτά υπόψη, αλλά η Κομισιόν διαπραγματεύτηκε μια νέα συμφωνία με τον Μάρκο χωρί να έχουν ακόμη διορθωθεί τα ασφάλματα του παλαιού συστήματο. Πρέπει τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει σοβαρά τις ευθύνες της και να αρχίσει να ερευνά πού γίνονται απάτες και να ζητήσει επίσης ε, επιστροφή των δασμών που δεν καταβλήθηκαν πριν γίνει η έγκριση, ε, η κύρωση αυτής της νέας συμφωνίας με το Μαρόκο. Δεν θέλουμε να μην υπογράφονται συμφωνίες, απλά οι συμφωνίες αυτές δεν θα πρέπει να πλήττουν ε, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Θα πρέπει επίσης οι κανόνες που έχουν υπογράφει στο πλαίσιο των συμφωνίων να τηρούνται. Σε σχέση με τη συμφωνία αυτή με το Μαρόκο, ο τομέας των αποκυρευτικών, ε, τι ζητάει ο κλάδος. Ζητάει εγγύηση να υπάρχει τήρηση των μέτρων τα οποία έχουν συμφωνηθεί και αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω της μεταρρύθμισης του καθεστώτος ε, υπολογισμού των τιμών εισόδου. Αν δεν υπάρξει νέο σύστημα τιμών εισόδου, δεν μπορούμε να έχουμε νέα συμφωνία με το Μαρόκο. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να κυρώσουμε τη συμφωνία που έχει ήδη κλείσει η Επιτροπή με το Μαρόκο. Επίση, είναι ευθύνη των κρατών μελών ο έλεγχο. Πρέπει να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερη οικονομική προσπάθεια, μεν, αλλά ε, ταυτόχρονα πρέπει να σα πω ότι εδώ και καιρό ζητούμε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα τελωνίων, όπω αυτό που υπάρχει στη ΣΥΠΑ, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την άποψη των Ισπανών παραγωγών οι οποίοι κατέθεσαν αυτή την καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών υπάρχει κίνδυνος που απορρέει από τις ε, ντομάτες του Μαρόκου και το πρόβλημα αφορά την τιμή εισόδου. Ε, Εμεί έχουμε διμερεί επαφέ με το Μαρόκο και στο πλαίσιο αυτών των επαφών καθορίσαμε την τιμή. Η Eurostat τον Δεκέμβρη του περασμένου έτου ε, εξήγαγε πάνω από 70.000 ντομάτε. Ε, πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που προβλέπει η ποσόστοση που έχει καθοριστεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Και αυτό οδήγησε σε πολύ μεγάλη ζημιά των Ευρωπαίων παραγωγών και μάλιστα δεν έχουμε συνυπολογίσει και του μη καταβληθέντε δασμού. Γι' αυτό λοιπόν σωστό είναι αυτό που λέγεται ότι πράγματι προέκυψαν παρατυπίες διότι έχουμε χαμηλότερες τιμές, εφαρμόζουμε χαμηλότερες τιμές από αυτές που ορίζονται στη συμφωνία και τούτο οδηγεί σε απώλεια εσόδων. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να υποβάλω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκ μέρους των υπολείπων μελών της Επιτροπής Αναφορών. Τι είδους μέτρα προβλέπετε και ποιο είναι το κόστος και η ζημιά που έχετε προϋπολογίσει τρεμό Μπαλθέλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον προηγούμενο Οκτώβριο είχα ε, υποβάλει προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τι διαφορέ μεταξύ ε, των στοιχείων που δίνονται από τι διάφορες υπηρεσίε ό,τι αφορά την εισαγωγή τομάτα από το Μαρόκο. Το 2008 περίπου 100.000 τόνοι μεταξύ γάμα τάξου και γύρω στα ήταν διαφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απαντήσει ότι πράγματι είχε εντοπίσει το πρόβλημα και το επέλει. Ήταν στην, σε εξέλιξη διαδικασία επίλυση. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον θα πετύχει η Κομισιόν αυτό που οι Ευρωπαϊκοί πολίτε και η Ευρωπαϊκή παραγωγή δικαιούνται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγουμε το όχι μόνο από το Μαρόκο, αλλά και από άλλε τρίτε χώρε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο οι διαπραγματεύσει να είναι δίκαιε προ όλου και να μην είναι σε βάρο του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Επίσης θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ελέγξουμε τι πραγματικά εισάγουμε από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίω ε, κάποια, ε, σε κάποια ευρωπαϊκά βόρεια λιμάνια. Πρέπει να είναι αποτελεσματική η συνοριακή έλεγχη, γιατί αλλιώς ο ευρωπαϊκός κλάδος Γεωργίας θα έχει πολύ δύσκολο μέλλον μπροστά του υπάρχουν απώλειες ε, στην ευρωπαϊκή παραγωγή ε, γεωργίας. Μάλλον αν υπάρξουν τέτοιες απώλειες θα είναι πολύ δύσκολο ε, να έχουμε εκ νέου παραγωγή ντομάτα στο έδαφο, αν υπάρχει πρόβλημα όλε αυτέ τι συμφωνίε, π.χ. με το Μαρόκο. Πρέπει να υπάρχει όμω δίκαιο ανταγωνισμό. Αυτό το δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε όμω την μη δίκαιη εφαρμογή κάποιων κανόνων ή που δεν ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για όλους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό, αλλά δεν θέλουμε να επηρεαστεί το εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υπέρ του ελευθέρου εμπορίου, αλλά υπό συμμετρικού όρου προστασία και ενημέρωση. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι, δεν είναι δίκαιο εμπόριο το ελεύθερο εμπόριο. Και ο ανταγωνισμό δεν είναι θεμητό ανταγωνισμό. Τέλο. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο, θα συμπεριληφθούν κάποιε ρήτρε για την αγορά εργασία, την κοινωνική διάσταση και το περιβάλλον στο Μαρόκο. Αν αυτό δεν συμβεί, ίσω έχουμε απώλειε ε, και στην ε, γεωργία και στον τομέα εφοδιασμού σε τρόφιμα. Ευχαριστώ. Κριστίνα, θέλει θέλεις για το Catch the Eye ή να μιλήσει ε, να απευθύνει τον τελευταίο μιλητή. Thank you, Mr. Ferreira. Ο κύριος Φερέιρα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τα αγροτικά προϊόντα για τα τρόφιμα με το Μαρόκο, με την Αίγυπτο ή το Ισραήλ, είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε πει ότι οι συμφωνίες αυτές θα πίεζαν προς τα κάτω τις τιμές των τροφίμων. Και αυτό είδαμε ιδιαίτερα στην Πορτογαλία όπου οι αγρότες έχουν όλο και, μεγαλύτερο πρόβλημα να διαθέσουν τα προϊόντα τους, μεσογειακά προϊόντα και λαχανικά και φρούτα, διότι οι... τα μεγάλα σούπερ μάρκετ αγοράζουν από άλλους Πάντοτε λέγαμε ότι η απελευθέρωση της παραγωγής τελικά θα ωφελούσε τις μεγάλες αγροτοβιομηχανίες προς ζημίαν των μικρών παραγωγών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες ως προς την τροφιμική μας ασφάλεια. Δυστυχώς είχαμε δίκιο. Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τους φόβους μας η Κομισιόν εδώ και χρόνια κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και δεν προασπίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γεωργών, των μικρομεσαίων ιδίως, γιατί αγνοεί, αγνόησε την έκθεση της Όλαφ όπου καταδικάζονταν οι ανομαλίες κατά τις εισαγωγές, οι ατασταλείς κατά τις εισαγωγές μαροκινής ντομάτας που οδήγησαν σε μείωση της τομάτης στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν αρνείται απλώς να εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπει η συμφωνία αλλά φροντίζει να συνάψει μία ακόμη πιο φιλελεύθερη που θυσιάζει τα συμφέροντα των μικροπαραγωγών προς όφελος των μεγαλύτερων. Πώς θα αποζημιωθούν οι μικροί. Μάτο Αλδοβέ, ευχαριστώ πολύ. Η παραγωγή από τις Κανάρες, τη Μούρθια, την Ανταλουσία, τη Βαλένθια, κοινοτική παραγωγή, παραγωγή τομάτας, ζητούν από την Κομισιόν να λάβει αποφασιστικά μέτρα έναντι μιας άδικης κατάστασης που δημιουργεί απάτες. Το είπατε κι εσείς. Χάρη στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαρόκο αποφελείται από μια τιμή εισόδου δεν θα πρέπει ε, να δούμε το 2007, ούτε στο, το 2010 τήρησε αυτή την τιμή εισόδου. Η τοματοπαραγωγή της Ισπανίας πρέπει να ανταγωνιστούν με τους Μαροκινούς, αλλά υπό διακριτικές ε, ε, συνθήκες και έτσι παίρνουν, αναλαμβάνουν πολύ ψηλότερα έξοδα παραγωγής λόγω των απαιτητικών κανόνων της Ένωσης για τα πρότυπα ποιότητα και ασφάλιση των τροφίμων, για τα εργατικά ζητήματα ή άλλες διατάξεις που δεν ισχύουν για τρίτες χώρες. Έτσι η δική μας παραγωγή που προσπαθούν, που ε, προσπαθούν να έχουν την κατάλληλη ποιότητα, αγωνίζονται για να σώσουν τις παραγωγές τους και τις καλλιεργίες τους. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι η Κομισιόν να μην ε, βλέπει την ε, μη εφαρμογή αυτού του καθεστώτος τιμής εισόδου, κάτι που ευνοεί και τις απάτες. Το είπε η Όλαφ. Η Κομισιόν όμως κοιτά από την άλλη πλευρά. Δεν επαρκεί δεν αρκεί να μα λέει η Κομισιόν ότι η επαγρύπνηση και επιτήρηση είναι αρμοδιότητα των κρατών μέλων. Γιατί αν δεν τηρούν τα κράτη-μέλη τι υποχρεώσει του, πρέπει να δράσει η Κομισιόν. Αυτό που δεν είναι ανεκτό είναι να καταπατώνται οι ε, όγκοι που πρέπει να εισαχθούν από το Μαρόκο χωρίς να καταβάλλονται οι δασμοί και να κάθεται σταυρωμένα χέρια κομισιών η οποία θέλει να εγκρίσει, εγκρίνει μια νέα συμφωνία συνέσης με το Μάροκο. Ας μην υπολογίζει τη δική μας έγκριση αν δεν τηρήσει τα δέοντα. Δεν θα πρέπει να κάνουν να τον ανταγωνισμό οι Μαροκινοί με τους Ισπανούς στοματοπαραγωγού. Καλό είναι να τηρούνται οι συμφωνίες, αλλά η υποχρέωσή σας είναι να προασπίσετε τα συμφέροντα των παραγωγών της Βαλένθια, της Ανδαλουσίας, ε, της ε, Μούρθια και όλων των άλλων περιοχών. Ευχαριστώ. Κάντε κάτι πριν είναι αργά. Αντρές Μπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Από το 2003 ζητούμε να αλλάξει ο κανονισμός για τις τιμές εισόδου. Ζήτησε το κοινοβούλιο μας αλλαγή, το ζήτησαν τα κράτη-μέλη, Ισπανία, Γαλλία, στηρίχθηκε αυτή η πρόταση από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Στόχος είναι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι ε, υπολογισμοί οι οποίοι δεν, ε, τελικά έχουν ως αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι τιμές εισόδου, να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και τελικά να εισπράττονται και μικρότερο, λιγότεροι δασμοί εισαγωγής. Αυτό βλάπτει τους ε, ο παραγωγούς απορροκυπευτικών. το άρθρο 5 του κανονισμού λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λογική εφαρμογή και λέει ότι ο με τον υπολογισμό τιμή εισόδου δεν καταβάλλονται κάποιοι πρόσθεσμοι. Λοιπόν, πρέπει η Κομισιόν να βρει μια λύση να δώσει μια απάντηση στο παραγωγικό σύστημα, αλλά να απαντήσει και στα κράτη. 16 χρόνια έχουν περάσει ότι ο μέας των απορροκυπευτικών στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στη Βαλένθια, στη Μούρφια, στην Ανδαλουσία επηρεάζεται, πλήττεται και θα πρέπει πλέον να υπάρξει κάποια λύση. Και πλήττονται και οι καταναλωτές. Ευχαριστώ. Δεκάστρο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η καταγγελία για την οποία συζητάμε σήμερα φτάνει σε κάποια μια στιγμή όπου η Επιτροπή Γεωργία και η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητούν για το νέο κεφάλαιο τη ε, Γεωργία για τη συμφωνία με το Μαρόκο. Η Όλαφ ε, μα διαβεβαιώνει ότι πράγματι υπήρξαν παρατυπίε όσον αφορά τον υπολογισμό δασμών για την εισαγωγή ντομάτα και ότι έχει προκύψει ζημιά για του Ευρωπαίου παραγωγού. Και οι ίδιοι παραγωγοί εκφράζουν την ανησυχία του ε, γιατί αυξάνεται αυξάνεται όλο και περισσότερο η εισαγωγή ντομάτας και οποροκυπευτικών και αυτό θα γίνει χειρότερα αν υπογραφεί η συμφωνία. Έχουμε λοιπόν αυτές τις διμερείς ε, συμφωνίες οι οποίες θυσιάζουν τη γεωργία προς όφελος άλλων βιομηχανικών συμφερόντων. Αυτό λοιπόν δεν <clears throat> είναι σωστό και θέλω να πω ότι σε μια κατάσταση οικονομικής, πολιτικής κρίσης σε όλη την περιοχή του Μαγκρέμ ε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιδείξουμε και κάποια λεγγύη στα πλαίσια της συμφωνίας που θα συναυθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως λένε και οι αναφέροντες από την ΦΕΠΕΞ, θα πρέπει η Κομισιόν να τροποποιήσει. Είναι μια αναφορά και της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών επίσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν κάποια άρθρα του κανονισμού. Επαναλαμβάνω να τροποποιήσει η Κομισιόν κάποια άρθρα του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά τον μέθοδο υπολογισμού τιμής εισόδου, πρέπει μία από τις τρεις μεθόδους ε, που λέγεται μέθοδος αφαίρεση, αυτή πρέπει να πάψει να ισχύει. Αυτό είναι σημαντικό, ε, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη, ότι οι ε, παραγωγή και οι εισαγωγέ επιλέγουν, οι εξαγωγέ μάλλον επιλέγουν αυτή η μέθοδο που του συμφέρει περισσότερο για να μην πληρώσουν του ε, δασμού. Τώρα που ε, έχουμε αυτή τη νέα συμφωνία με το Μαρόκο που είναι προ έγκριση, θα πρέπει η Κομισιόν μία ε, για πάντα πλέον να διορθώσει το σύστημα. Εμείς σήμερα για μια ακόμη φορά επιμένουμε. Η καλή λειτουργία των τιμών εισόδου είναι ένα λογικό αντιστάθμα που μπορούν να αναμένουν οι παραγωγοί μας ε, όταν θα τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Διαδικασία δια. Λαβία. Signor Presidente, signor Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εγώ πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση μετά από την καταγγελία που κατέθεσε η FedEx είναι μια ε, συζήτηση ιδιαίτερα επίκαιρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο παράλληλα συζητάει και την εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο. Η καταγγελία είναι σαφές ότι επισημαίνει ένα πρόβλημα ε, επί του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ζητάει κατηγορηματικά αυτήν την απάντηση από την Επιτροπή πριν προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να πληρώνουμε, να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί αυτή την κατάσταση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προστατεύσουμε τους δικούς μας, τους γεωργούς και τούτο όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή της ντομάτας αλλά γενικότερα όσον αφορά την παραγωγή των οπωροκυπευτικών, μια παραγωγή που θα πληγεί σημαντικά εάν πράγματι ανοίξει χωρίς εξαιρέσεις το εμπόριο. Ο κύριος Παντσέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κατανοώ βέβαια την κριτική που ασκήθηκε σήμερα το πρωί όσον αφορά την καταγγελία που κατατέθηκε. Νομίζω ότι πράγματι ε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά σχετικά με αυτή τη συμφωνία για τα απορροκυπευτικά με το Μαρόκο έτσι ώστε η συμφωνία να τύχει συνένεση. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει αφενό να καλύπτει τι ανάγκε ισορροπία, να μην αντιμετωπίσουν πάρα πολλέ δυσκολίε η Ευρωπαϊκή παραγωγή, από την άλλη όμω να υπάρχουν και σαφεί και διαφανεί κανόνε για τον ανταγωνισμό στην αγορά αγορά γεωργίας. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Έτσι λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει τις σωστές λύσεις χωρίς να αγνοεί τα συμφέροντα των παραγωγών όμως παράλληλα και χωρίς να αγνοεί ότι πρέπει να έχουμε μια γενναιόδορη πολιτική απέναντι στο Μαρόκο κυρίως λαμβάνω υπόψη όλα αυτά που διαδραματίζονται στο Μαγκρέπ. Πρέπει λοιπόν να τα κατανοήσουμε όλα αυτά και εγώ ε, δεν νομίζω ότι ότι τελικά αντί να εισάγουμε ε, την ντομάτα να εισάγουμε και όλα τα άλλα παραπροϊόντα της ντομάτας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να εξευρεθεί μια νέα και σωστή ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Ο κύριος Ρομέρα. Ευχαριστώ. Ε, το business as usual ε, δεν έχει δώσει πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσματα και τώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδίω σε σχέση με τα όσα γίνονται στο Μαγκρέμπ σήμερα. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε, δεν θα ήταν λογικό να συνεχίσουμε με αυτή τη ε, συμφωνία. Εγώ είμαι εισηγητής ε, για τη σχετική έκθεση στην Επιτροπή Αλίας. Θα πρέπει να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Να πούμε ξεκάθαρα ότι να ζητάμε η τομάτα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που εισάγεται να εισάγεται υπό τις ίδιες συνθήκες ε, με ε, τις οποίες, πρέπει να πληρούν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και αν δεν ε, υπάρχει σχετική εγγύηση πρέπει, οφείλουμε και ελπίζω να το κάνει και το Κοινοβούλιο να το ξαναδούμε όλο το, το πλαίσιο δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική προστατευτισμού, αλλά τουλάχιστον δικαιοσύνη, εμπορική δικαιοσύνη. Και θα πρέπει να δούμε μέσα σε ποιο πλαίσιο μπορούμε να δράσουμε και να δράσουμε τον πλέον υπεύθυνο τρόπο. Ευχαριστώ. Γκουτιέρεθ Κορτίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατανοούν ε, το πρόβλημα της Μεσογείου, την Ισπανική αντιπροσωπεία που καταλαβαίνουν ότι Κανάρις, Αλμερία, η Μούρθια, η Βαλένθια και απογοητεύονται διότι δεν ε, πληρείται τις συμφωνίες η Κομισιόν και δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να δεχόμεθα μετανάστες από τον υποσαχάριο Αφρική, από το Μαρόκο και να είμαστε τελικά ο κυματοθράφστης μπροστά στην κρίση. Βλέποντας ότι υπάρχουν δεινές οικονομικές συνθήκες, έχουμε άτομα τα οποία έρχονται για να, να δουλέψουν στις χώρες μας και να στείλουν κάποια χρήματα στις οικογένειές τους. Ενώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ε, στις χώρες μας τελικά. Δεν έχετε σκεφτεί νομίζω από πλευρά Κομισιόν πώς θα προασπίσετε τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν πρέπει να ανοίξετε ε, σε αυτή τη, την πόρτα σε αυτή την πολιτική που έχει ω αποτέλεσμα να εισάγονται προϊόντα με πολύ αμφίβολες φυτογειονομικές ε, ιδιότητες. Ευχαριστώ. Γεια. Herr Präsident, der Europäische ε, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ιστορική Αγορά συστήθηκε για να ανταποκριθεί καλύτερα στην προστασία του καταναλωτή. Ο καταναλωτή έχει δικαίωμα στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αγοράζει υγιή προϊόντα. Το άνοιγμα τη αγορά ε, αυτό όμω συνεπάγεται και εισαγόμενε, ελεγχόμενε εισαγόμενε ποσοστώσει. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα εξή. Πρώτον, οι εισαγόμενε ποσότητε πρέπει σαφώ να ελέγχονται. Αυτό αφορά κυρίω και πάνω απ' όλα ε, το ποσοτικό στοιχείο. Δεύτερον, όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, και αυτή πρέπει να ελέγχεται αυτό αφορά ε, και τις προδιαγραφές παραγωγής και τρίτον οι επιπτώσεις στους ε, γεωργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, να γίνονται δοσοληψίες και αγορές εις βάρος τρίτων αυτό σημαίνει κυρίως αγορές προς όφελος βιομηχανίας και εις βάρος των γεωργών αυτό πρέπει να αποφεύγεται γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει πολύ προσεκτικά τη συμφωνία, την επικείμενη συμφωνία με το Μαρόκο και μόνο εφόσον πράξει Γι' αυτό, τότε να προχωρήσει στη σύναψή της. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ισπανούς παραγωγούς οι οποίοι μας υπέβαλαν την αναφορά αυτή που είναι πολύ επίκαιρη. Γιατί εδώ και μήνες στο Κοινοβούλιο Έχουμε προσπαθήσει να επιστήσουμε στην προσοχή των κίνδυνο που ε, συνεπάγονται κάποιες διμερείς συμφωνίες. Φυσικά και μας ευαισθητοποιεί το ζήτημα του Μαρόκου και γνωρίζουμε ότι ο καθορισμός το να τους αναγκάσουμε τους Μαροκινούς να μείνουν στη χώρα τους είναι η καλύτερη λύση και ε, θα μας αποτρέψουν από μελλοντικά προβλήματα μετανάστευσης, αλλά μάλλον αν φτιάξουμε τα πράγματα στη χώρα του Μαρόκου. Αλλά το να εγκρίνουμε και να επικυρώνουμε κάποιες καταστάσεις, όπως βλέπουμε και μέσω των εκθέσεων της Όλαφ, τελικά η λύση που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι κατάλληλη. Και θέλω να σας επισημάνω και έναν άλλο κίνδυνο. Μα λέτε ότι οι συμφωνίε που θα επαναδιαπραγματευτεί θα έχουν σαν να στηρίξουμε του Μαροκινού παραγωγού. Μα και ποιου Μαροκινού παραγωγού μιλάμε οι είναι από μεγάλες γεωργοδιατροφικέ αλυσίδες που έχουν εγκαταστήσει στο Μαρόκο μεγάλες, τεράστιες εκμεταλλεύσεις. Δεν είναι η μικρό παραγωγή από το Μαρόκο αυτή που ωφελούνται από συμφωνίες μας, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υπό αποδεκτούς για την ευρωπαϊκή αγορά όρους. Γι' αυτό λοιπόν να μην αυτά πατώμεθα, αλλά και να μην απογοητεύουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό ζητώ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την άδειά σας να σας αναφέρω μερικά στατιστικά στοιχεία για να απαντήσω σε αυτά που είπαν ορισμένοι συνάδελφοι. Ορισμένοι βουλευτές από 185.000 τόνους περάσαμε σε 295.000 295.000 και τα νοπά προϊόντα αυξήθηκαν παντού από 233.455 και το μερίδιο του Μαρόκου έπεσε από το 76% σε 59. Μάλιστα, θα έλεγα ότι οι ντομάτες που παρουσιάζονται στον κόσμο είναι 80 εκατομμύρια τόνοι εξών 16 περίπου για κατανάλωση άμεση. Τώρα για τη νέα συμφωνία με το Μαρόκο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι συμφωνία πολύ λίγο και πολύ ισορροπημένη και η Κομισιόν θα προσέξει ιδιαίτερα να γίνουν σεβαστοί όλοι οι όροι και ρήτρε και κανόνες. Οι καινούργιες ποσότητες που προβλέπει η ποσόστοση προβλέπονται από τους κανόνες ακριβώς αυτούς. αυτούς. Οι 52.000 πρόσθετοι τόνοι με τους τόνους αυτούς φτάνουμε τις 180.000 δηλαδή την ποσόστοση. Δεν ξεπερνάμε την ποσόστοση. Τώρα αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα, μια άλλη πτυχή του προβλήματος. Μας κατηγορούν ότι μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτή η κατηγορία όμως είναι άδικη και λανθασμένη. Μία μόνο περίπτωση σημειώθηκε ατασταλίας και η Όλαφ την ανέφερε δεόντως μετά από την νομισμένη έρευνα. Έγινε κάποια δίκη στη Γαλλία και επιστράφηκε ένα τμήμα του ποσού που είχε τύχει κατάχρησης. Όσο για τους υπόλοιπους κανόνες να είστε βέβαιοι ότι εμείς σεβόμαστε όλες τις προδιαγραφές αυστηρότατα για όλες τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών και οποροκυπεφουτικών γενικότερα στην Ένωση. Κατανοώ ότι, μπορεί, ότι οι ευρωβουλευτές θέλουν να το προσέξουν ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι και οι αγρότες, και οι αγρότες πρέπει να προσέχουν με τον ίδιο τρόπο όσοι έχουν στοιχεία για απάτη να τα υποβάλουν στην Κομισιόν και θα κάνει τα δέοντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Διάλειμμα μέχρι τα 12.